καλύτερη στο μέλλον συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Η συζήτηση τελείωσε. Η ψηφοφορία ε, θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η έκθεση της ε, κυρίας Γκαρσία Πέρετ «Συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών». Θα λάβει τον λόγο η κυρία εισηγήτρια. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ κυρία Πέρετ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι περίπου το 70% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 83% της, ε, του δραστήριου πληθυσμού από πλευράς γυναικών είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Γι' αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας η εργασία που αναπτύχθηκε σε σχέση με την ε, Επιτροπή Ισότητας για αυτή την έκθεση. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας για το έργο που έγινε με τις τροπολογίες και τη διαπραγμάτευση επ' αυτών μεταξύ συναδέλφων γυναικών και ανδρών που έδωσαν δυνατότητα να επανεπεξεργαστούμε την αρχική έκθεση. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε αυτήν την έκθεση θέματα όπως τον επισφαλή χαρακτήρα εργασίας, τα στερεότυπα, το ψηφιακό χάσμα, την ε, συμφιλίωση και συνδιαλλαγή, τις νέες ε, τεχνολογίες, ε, θέματα που έχουν τεράστια σημασία για την ισότητα και για την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό όμως να γίνεται αναφορά σε κάποια σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν και αυτά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στους κόλπους της Επιτροπής μας σε σχέση με την ελαστικότητα αληθεύει ότι η ελαστικότητα, η εργασιακή ελαστικότητα κάποιες χρονικές στιγμές μπορεί να ευνοήσει την ένταξη των γυναικών στην εργασία και την δυνατότητα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η ελαστικότητα αυτή δεν μπορεί να είναι εις βάρος των γυναικών. Να καθορίζει ο ίδιος ο, ο επιχειρηματίας τους όρους και να, ο ίδιος να επιβάλλει την ε, ελαστική απασχόληση. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ε, οικογενειακής ζωής για τις, γυναίκες, Ένα άλλο θέμα που εξετάσαμε σε αυτήν την έκθεση είναι οι συμβάσεις ε, περιορισμένου χρόνου και μερικής εργασίας που ε, είναι θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Όμως ως δυνατότητα πρέπει να προσφέρεται. Δυνατότητα που θα είναι στην ελεύθερη επιλογή των γυναικών, των ιδίων να δουν αν θα τις υιοθετήσουν ή όχι στην εργασιακή αγορά. Να μην ξεχνάμε ότι όταν κάνουμε λόγο για συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κάνουμε λόγο για υποχρέωση, υπευθυνότητα ανδρών και γυναικών και δεν μπορεί αυτό να γίνεται εις βάρος των γυναικών, να πληρώνουν τα σπασμένα οι γυναίκες όπως ε, όταν εκείνες ασχολούνται αποκλειστικά με την μέρημνα και φροντίδα των παιδιών και των υπερήλικων στην οικογένεια. Θελήσαμε να δώσουμε μια συνιστόσα για τη σπουδαιότητα που έχουν οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, τα εξαρτώμενα άτομα. 80% των όσων προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες σήμερα είναι γυναίκες. Χρειαζόμαστε κοινωνικές υπηρεσίες αναβαθμισμένες και δωρεάν και να μην ε, αποσυναρμολογήσουμε το κοινωνικό κράτος όπως συμβαίνει σε πολλές ε, χώρες σήμερα με την κατάργηση κοινωνικών υπηρεσιών και θα πρέπει να μπορέσουμε να εντάξουμε τις γυναίκες μέσα σε αυτό το πλαίσιο σε ένα πλαίσιο ισότητας στην αγορά εργασίας. Θέλουμε επίσης να θίξουμε ένα θέμα όπως είναι το χάσμα το μισθολογικό, οι διαφορές μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών. Υπάρχει αυτό το χάσμα το μισθολογικό εις βάρος των γυναικών. Έχουμε μερική απασχόληση για τις γυναίκες, επισφαλή απασχόληση για τις γυναίκες που οδηγούν όχι μόνο στο να υπάρχει μισθολογική διαφορά σε σχέση με τους μισθούς που καταβάλλονται στις γυναίκες, αλλά επίσης να βλέπουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο και το γεγονός ότι τα δικαιώματα σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τις γυναίκες αυτές να είναι πολύ μικρότερα από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ανδρών. Το μισθολογικό χάσμα, το μισθολογικό αυτό κενό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να εργαστούν τα κράτη-μέλη ώστε να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα όσα αναφέρονται στις ε, επιθεωρήσεις εργασίας για τους όρους απασχόλησης και την επίτευξη των πολιτικών απασχόλησης από πλευρά των επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αμελήσουμε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Κάνουμε επίση αναφορά στην ανάγκη του να επανεξεταστεί το θέμα όσον αφορά τις, ε, την οδηγία για την γονεϊκή άδεια είναι μια, ένα αίτημα που από το Κοινοβούλιο διατυπώνουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο για γονεϊκή άδεια για τις γυναίκες, αλλά είναι σημαντική επίσης υπόθεση και η, γονεϊκή άδεια και για τους ε, άνδρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή η οικονομική κρίση να επιδεινώσει την ε, εργασιακή αγορά και τους όρους απασχόλησης των γυναικών. Διότι στο τέλος τέλος θα πλήττονται εκείνα τα άτομα τα οποία θα έχουν περισσότερες δυσκολίες και θα είναι πιο ευάλωτα και όλα αυτά θα τα πληρώσουν ως σπασμένα, τα σπασμένα οι γυναίκες. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας και να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Τσιρέσκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή που αναφέρεται στο ρόλο των γυναικών στον τομέα της ε, εργασίας, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, αν και η απασχόληση των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών είναι αρκετά υψηλή. Οι γυναίκες υφίστανται βέβαια πάρα πολλά προβλήματα, πολλές φορές έχουν προβλήματα κατάρτισης, έχουν μειωμένε μειωμένες απολαβές για την ίδια εργασία με τους άνδρες και πολλές φορές εργάζονται με μειωμένο ωράριο και πληρώνονται αντίστοιχα φυσικά. Προσπαθούν να συνδυάσουν την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές Γι' αυτό ζητάμε να υπάρχουν υποδομές για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων. Και οι εργοδότες και οι οργανώσεις των εργαζομένων θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε η εργασία των γυναικών να έχει την ίδια αξία με την εργασία των ανδρών. Η κυρία Βέτμαν. Είναι θλιβερό γεγονός ακόμα, αλλά αληθεύει. Οι γυναίκες 16,4% μικρό, χαμηλότερους μισθούς έχουν από τους μισθούς των ανδρών. Και στη χώρα μου οι γυναίκες 60% έχουν μόνο από τον ε, μισθό των ε, ανδρών. Υπάρχει λοιπόν διαφορετική ε, αναφορά σε σχέση με τις γυναίκες και βλέπουμε ότι πολύ λίγες γυναίκες στα, σε ηγετικά κλιμάκια είχαν προχωρήσει. Οι γυναίκες θα πρέπει να προσελκυστούν σε αυτές τις θέσεις όπως και οι άνδρες. Όμως θα πρέπει να συμφιλειωθεί η επαγγελματική δραστηριότητα με την οικογενειακή ζωή και να μπορέσουν να υπάρξουν δυνατότητες κατάτησης και επιμόρφωσης για τις γυναίκες ώστε να πορεθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Πένιοβα στη συνέχεια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον τομέα των υπηρεσιών σχεδόν 70% βλέπουμε ότι σημειώνεται απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών είναι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των απασχολούμενων γυναίκες. Εργάζονται ποσοστιαία περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες στον τομέα των υπηρεσιών. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Υπάρχουν ε, στερεότυπα, άκαμπτα στερεότυπα που έχουν βαθιές ρίζες φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες δουλειές, κάποιες εργασίες οι οποίες είναι εντός εισαγωγικών γυναικείες, άλλες που είναι ανδρικές πάλι εντός εισαγωγικών. Όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα στις α, ιδεολειπτικές προσεγγίσεις ότι η θέση των γυναικών είναι στο σπίτι και ούτως ή άλλως είναι χαμηλόμιστες οι γυναίκες οι γυναίκες 17% κατά μέσο όρο ε, έχουν χαμηλότερους μισθούς από ότι οι άνδρες Επίσης 80% όλων των χαμηλότερων μισθοδοτούμενων στην Ένωση είναι γυναίκες. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κάτι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, 83,1% των γυναικών που απασχολούνται απασχολούνται στο τομέα των υπηρεσιών και μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι επικεντρώνεται κυρίως σε ορισμένους τομείς όπως τις φροντίδες, διαμετζαγώγησης, ε, του μάρκετινγκ, ε, της ε, εκπαίδευσης και αυτό έχει απαραίτητα με βάση τα στερεότυπα τα οποία προβάλλει η έκθεση. Υπάρχουν υποθέσεις ότι ιδιαίτερε είναι οι ικανότητες αυτές των γυναικών όπως τη διαμεσολάβηση ή του μάρκετινγκ που τους επιτρέπουν να δουλεύουν στους τομείς αυτούς και ότι μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα από ότι οι άρενες συναδελφοί τους στους τομείς αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αντί να απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένο φύλλο για το κάθε επάγγελμα να αναπτύσσουμε επαγγέλματα για ανθρώπους και να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα οδηγούν στη φτώχεια και ε, την υποβάθμιση του επέδου ζωή. Ε, μία μπλε κάρτα, κύριε Μπερμάιερ, στη δεθμένος να τη δεχθείτε. Βεβαίως, έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπερμάιερ αν θεωρεί ότι οι γυναίκε ε, θα μπορούσαν να είναι καλύτερε ω πολιτικοί. Θεωρείτε ότι οι γυναίκε πολιτικοί μπορεί να είναι ικανέ. Ε, δεδομένου ότι έχουμε τόσο μεγάλες ικανότητες διαμεσολάβηση, παιδεία, διαπαιδαγώγηση κτλ. που χρειάζονται τόσο πολύ στην ε, πολιτική. Κύριε Μπερμάιερ, θα απαντήσετε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είχα πει εξ αρχής ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερη δυνατότητα ενσυναίσθησης περισσότερο από ότι οι άντρες και γι' αυτό νομίζω ότι και στην πολιτική αλλά και σε ηγετικέ θέσει, όπως άλλωστε ακούστηκε και νωρίτερα, είναι σημαντικό χωρίς όμως ποσοστώσεις να υπάρχουν πολλές γυναίκες. Πιστεύω ότι η λύση με τις ποσοστώσεις θα ήταν μια ασφαλμένη λύση, μια ασφαλμένη προσέγγιση. Αλλά ασφαλώς θα πρέπει, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, να υπάρχει ισότιμη αμοιβή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μια ακόμη μπλε κάρτα για εσάς από την κυρία Τσίσκοβα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να, απαντήσω, να τα αντιδράσω μάλλον σε κάτι που ακούστηκε τώρα μόλις. Για το κατά πόσον χρειαζόμαστε περισσότερους ε, άνδρες ή έχουμε μάλλον περισσότερους άνδρες ε, δασκάλους ε, και ερωτώ γιατί να μην υπάρχουν δάσκαλοι και βέβαια νηπιαγωγοί άνδρες δεν έχουν να κάνουν και, αυτά με και αυτοί με παιδιά. Δεν χρειάζονται παιδιά άντρες ε, στην θέση αυτή. Εγώ βλέπω από την εμπειρία μου ότι υπάρχουν αρκετοί νηπιαγωγοί και δάσκαλοι άντρες και είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η κάλυψη και από τα δύο φύλλα. Ο κύριος Σόμπερμαϊερ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπα, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει κανείς να υποχρεωθεί να το πράξει. Αν υπάρχουν και περισσότεροι άντρες που ενθουσιάζονται για αυτά τα επαγγέλματα, βεβαίως και είναι πολύ σωστό πολύ καλό. Δεν χρειάζεται όμως να υπογραμμίσω ακόμη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθύνονται τα επαγγέλματα σε ανθρώπους, είτε πρόκειται για φροντίδα, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Εάν ένα επάγγελμα αποκτήσει καλύτερη εικόνα στο κοινό, εάν θεωρηθεί δηλαδή πιο ελκυστικό, αν έχει και καλύτερη αμοιβή, ασφαλώ και άνδρες και γυναίκες θα προσελκύσει. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Μπασέσκου τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν ταυτόσιμες συνθήκες και όρους απασχόλησης. Όμως σε πολλές χώρες υπάρχουν διαφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση και στους μισθούς φυσικά. Και έτσι θα πρέπει να πούμε ότι το 2010 μόνο ένα από τα επτά μέλη των ε, συμβουλίων, διαχειριστικών συμβουλίων των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ένα από κάθε επτά ήταν γυναίκα και γι' αυτό θα πρέπει να προσπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών και στο αστικό τομέα. Οι όροι και ε, προϋποθέσεις απασχόλησης των γυναικών στις υπηρεσίες πρέπει να ε, είναι συμβατές με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και σε σχέση με τον σεβασμό των ε, βασικών αρχών για την απασχόληση και πρέπει να μεριμνούν τα κράτη-μέλη για την τήρηση αυτών των αρχών. Ευχαριστώ. Κυρία Ζαμπόσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα αυτών. Χρειαζόμαστε στα επαγγέλματα του ιατρού, του δασκάλου, πολύ περισσότερο προσωπικό. γυναίκες επιτοπλίστων είναι στο χώρο της δασκαλίας, ενώ αντίθετα στι διευθυντικέ θέσει είναι πολύ λιγότερε από ότι οι άντρες ή γυναίκες στις επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουν οι γυναίκες να συγκεράσουν τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο. Αυτό ισχύει φυσικά για, το, για τη γυναίκα όσο και για τον άντρα. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί απασχόληση για τα τρίτα τέταρτα των γυναικών όπως και των ανδρών και πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, ε, κάλυψη και υποδοχή και για τα παιδιά στα σχολεία. Οι γυναίκες οι οποίες όμως έχουν θελοντικά επιλέξει να μείνουν στην οικογένεια και να φροντίσουν για τα παιδιά τους θα πρέπει να, έχουν να τύχουν και, αυτή τις ίδιες, και αυτές τις ίδιες προσοχές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Τσέσκοβα, υπάρχουν ακόμη επαγγέλματα στα οποία υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκε σχέση με του άντρε και αυτό έχει να κάνει με τα στερεότυπα τα οποία έχουν επικρατήσει στις κοινωνίε μα. Συμφωνώ ότι οι γυναίκες επιτοπλίστων έχουν χαμηλότερες αμοιβέ και αντιμετωπίζουν όχι μόνο οριζόντια αλλά και κατακόρυφη διάκρισης βάρος τους στον χώρο της ε, ε, επαγγελματικής αδειοδρομίας. Χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν οι γυναίκες σε θέσεις με περισσότερο κύρος. Θέσεις ή επαγγέλματα όπως αυτό της φροντίδας την χάνουν ιδιαίτερης, ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία αναντικατάστατα είναι και χωρίς βέβαια να θέλω υπερβολικές ρυθμίσεις θεωρώ ότι θα πρέπει όπως είπαν και αρκετοί συνάδελφοι, να υπάρξουν ρυθμίσεις και για τον ευέλικτο τρόπο εργασίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ε, θα καταθέτει νέε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την απελευθέρωση, η τέλεια απελευθέρωση αυτού του τομέα, ε, παραδείγματι στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν κατοίκων Βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις ε, που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που όμως δεν είναι σε θέση να ε, υπαχθούν στις ρυθμίσεις οι οποίες ε, προτείνονται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μιράντα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, <clears throat> συγχαρητήρια για αυτή την έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Οι περισσότερε γυναίκε απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, όμω και το μεγαλύτερο μέρο των γυναικών έχουν επισφαλή εργασία προσωρινή και επισφαλή μερική εργασία υπό ε, χαμηλά αμοιβόμενη εργασία, μαύρη παραεργασία, πολλές φορές εις βάρος τους. Δεν εξυπηρετεί τις γυναίκες να τους δίνουν δουλειά με την ελαστικότητα και μάλιστα λέγοντας ότι υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις σε κάποια κράτη-μέλη που όπως στην Ισπανία ε, έχουμε την ε, ε, επιλογή της μερικής απασχόλησης και της ελαστικής απασχόλησης. Θέλουμε να έχουν επαρκή προστασία στην τομέα των υπηρεσιών οι γυναίκες. Για μια παρέμβαση από την κυρία Τίκαο. Θα θέλαμε να πω ότι 83,1% ε, το, ως ποσοστό των γυναικών εργάζεται στις υπηρεσίες. Ωστόσο το 78% του συνόλου της απασχόλησης ε, είναι θέσεις που ε, καταλαμβάνουν οι γυναίκες. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν μια στρατηγική με εξειδικευμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς όροι απασχόλησης των γυναικών και με, και με βάση τις συμβάσεις τους κιόλας. Ο αριθμός των γυναικών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο διαδίκτυο αυξάνεται. Πράγμα το οποίο όμως βλέπουμε ότι παρόλη την ε, ε, ανώτερη ε, μόρφωση των γυναικών υπάρχουν προβλήματα στο να διοχετευτούν στις, στις θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν επιμόρφωση και κατάρτιση στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε στις τεχνολογίες της ενημέρωσης και της πληροφόρησης να μπορούν να βρουν ικανοποιητική απασχόληση απασχόληση γυναίκες παράλληλα με τις ε, υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε το Καρστιά και ακούμε τώρα τον κύριο Νταλή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, εξαιρετούμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Γκαρσία Πέρες για την έκθεσή τη για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία δίνει μια ε, ευρία επισκόπηση, αλλά ζωφερή εικόνα, την οποία συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, πολύ σπάνια έχουν ηγετικέ θέσει οι γυναίκε και λίγε είναι ευκαιρίε για, για επαγγελματική αναρρίχηση. Δύσκολε συνθήκε ε, συγκερασμού του οικογενειακού με τον επαγγελματικού βίου και πολλές δυσκολίε. Η δε ύπαρξη παιδιών πολύ συχνά ε, κάμπτει σημαντικά τις προοπτικές για, για επαγγελματική ανάδειξη των γυναικών. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί μια απόφαση για απόκτηση παιδιού δεν μπορεί να αποτελεί φραγμό στην επαγγελματική σταδιοδρομία μια γυναίκα. Η υποεκπροσώπηση στου χώρου λήψη αποφάσεων, οι διάφοροι φραγμοί στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών έχει μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να μην υπάρχει συγκεκριμένο στόχο για ποσοστά ή ποσοστώσει αποσχόληση γυναικών σε ηγετικέ θέσει. Στη στρατηγική του 2007 αναφέρεται ότι ένα από το 27 της, της 100 για τις ηγετικές θέσεις ε, στην μεσαία ομάδα ηλικίας πρέπει να επιδιωχθεί. Και επίσης πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της στόχιας κατά 20 τουλάχιστον εκατομμύρια, που βέβαια μόνο με την καλύτερη συμπερίληψη των γυναικών στα προγράμματα για την καταπολέμηση της στόχιας μπορεί να επιτευχθεί. Δεύτερον, τα θέματα της ισότητας των φύλων, τα θέματα τα σχετικά με τον φύλων είχαν συζητηθεί και στην ενισχυμένη συνεργασία. Στο πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο εξάλλου αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να προταθούν λύσεις μείγματος πολιτικής για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και των λόγων που οδηγούν σε αυτό το 2011-2012 συστάσεις για ε, ορισμένα κράτη-μέλη εξεδόθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που και επικεντρώνονταν σε, ε, στην ανάγκη για παροχή απαραίτητων και ουσιοδών υπηρεσιών ώστε να υποφελούνται από τις εκτόσεις φόρων, να βοηθούνται οι γυναίκες για γενικότερα για την αντιμετώπιση του χάσματος ε, των φύλων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει βέβαια πρόοδου, σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ε, καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, καλεί τα κράτη-μέλη για πιο αποτελεσματική δράση στον τομέα αυτών θεωρώντας ότι η ισότιμη μεταχείριση για τις γυναίκες που χαρακτηρίζει πολλές από τις πολιτικές μας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για τη βελτίωση των συνδικών στην κοινωνία. Οι προτεραιότητες για τη στρατηγική για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που αναφέρεται σε δράσεις οριζόντιες για όλες τις γυναίκες, η αντιμετώπιση της διαφοράς της αμοιβέ, παραδείγματι, ε, είναι πολύ σημαντικό, στοιχείο. Πρέπει να αναστηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν και να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια έκθεση για την υλοποίηση της ε, οδηγίας της για την ίση, για την αμοιβή και τώρα προβλέπει μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τα ζητήματα αυτά της ισότητας και ιδιαίτερα της διαφοράς της αμοιβέ, κατάρτιση, βέλτιστες πρακτικές για και από επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν ήδη από το φθινόπωρο και επιπλέον σημειώνεται για άλλη μια φορά είχε εορτάζεται το 2013 η Ευρωπαϊκή ημέρα για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και γνωρίζετε πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών στον επιχειρησιακό χώρο με άνησες ακόμη εξελίξεις και προόδους θεωρούμε ότι είναι, θα, είναι απαραίτητο ίσως να προχωρήσουμε σε επιπλέον μέτρα. Επίσης θα ήθελα για την απασχόληση να επισημάνω ότι η ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι κύριος στόχος. Καλούμε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για την απασχόληση, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα επικεντρωνόμενα στη δημιουργία θέσεων εργασίας με τη χρήση και των ευρωτικών ταμείων και άλλων κονδυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιοποίηση κάθε δυνατής ε, ευκαιρίας και στρατηγικές για καλή απασχόληση μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό πλαίσιο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των γυναικών εργαζομένων σε σχέση δε με την τομεακή προσέγγιση του πακέτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει, προωθεί λευκές, πράσινες σταδιοδρομίες αλλά και σταδιοδρομίες στον χώρο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Τρίτον, η απασχόληση είναι καλύτερη εγγύηση για την αποφυγή της ανεργίας και του αποκλεισμού από την κοινωνία. Στην ε, τρέχουσα οικονομική δυσπραγία θα πρέπει η κοινωνική ενσωμάτωση να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να ενισχύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της επεξεργασίας πολιτικών απασχόλησης ώστε να λάβουν υπόψη, να, να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις και να βοηθήσουν τις γυναίκες να ενταχθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι οι διατάξει αυτές θα φέρουν πραγματικέ αλλαγές και θα κλείσουν το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα η σε διάταξη προβλέπει την ε, συζήτηση της εκθέσεως του κύριου Τριανταφυλλίδη, ενίσχυση της αλληλεγγύης